Liebe Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό είναι να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής μας και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκριση αυτής. Υπάρχουν διαφωνίες, αντιρρήσεις, ενστάσεις ως προς την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν τέτοιες αντιρρήσεις, επομένως εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη ως έχει. Δεύτερο θέμα, έγκριση των πρακτικών. Τα σχέδια των πρακτικών των συνεδριάσεων της 11ης Ιουλίου και της 4ης Σεπτεμβρίου βρίσκονται στα έγγραφά σας. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις να κάνετε για τα πρακτικά. Όχι. Γι' αυτό και προτείνω, ως συνήθως, να θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά εφόσον δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ενστάσεις έως το τέλος της ε, συνεδρίασής μας. Και φαίνεται να συμφωνείτε όλοι. Πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Υπάρχει σήμερα διερμηνία στις εξής γλώσσες γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Επίσης, ως συνήθως, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο και αποφάσεις συντονιστών 4 Σεπτεμβρίου. Λάβατε τις αποφάσεις αυτές στις 5 Σεπτεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχουν εγκριθεί καθώς έως την προθεσμία της 7 Σεπτεμβρίου δεν είχαν υποβληθεί αντιρρήσεις. Επομένως έχουν εγκριθεί και αυτές οι αποφάσεις των συντονιστών. Επόμενο θέμα ψηφοφορίε. Δύο είναι τα θέματα που θα τεθούν σε ψηφοφορία σήμερα. Δύο σχέδια γνωμοδοτήσεων. Πρώτον, έκθεση πρωτοβουλίας για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017, ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια ένωση της δημοκρατικής αλλαγής. Καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Αναφορών η Κριστίνα Μπάτσκα είναι δική μας εισηγήτρια. Ε, Κριστίνα, προς του, πέρασουμε στην πληροφορία, θέλεις να λάβεις το λόγο. Όχι. Επομένως μπορούμε να περάσουμε απευθείας στην ε, ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να βεβαιωθούμε. Ψηφίζουμε λοιπόν επί της τροπολογίας 10 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Okay. Geschlossen. Πέρασε Σαφής ήταν η διαφορά. 15 υπέρ, 3 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ,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 αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39. Όχι, εντάξει, ωραία. Θέλετε να ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. ψηφίσουμε για την τροπολογία 38. Ψηφίστε παρακαλώ. 38. 38. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. 15 υπέρ, 9 κατά, μία ε, αποχή εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται.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 ναι, Κριστίνα, παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θέλω να πάρω το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις, ευχαριστούμε τη γραμματεία, όλους τους βοηθούς. Πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά που ανέλαβα ε, τη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ και εγώ, Κριστίνα για τη δουλειά αυτή. Ήταν μια έκθεση που πραγματικά ε, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και έτσι περνάμε στην επόμενη συνεδρίαση έκθεση πρωτοβουλίας εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ε, ε, αναπηρία Καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή απασχόληση. Δική μας ε, η συγκέντρια είναι η Τζούλι Βόρτ. Θε να πεις κάτι Τζούλι? Όχι. Οπόμενο μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, διερμηνία προς τα αγγλικά από ό,τι με ενημερώνουν. Οκ. Alles klar. Wunderbar. Το λύσαμε. Τέλεια. Θέλεις να πεις κάτι Julie Ward? Όχι. Ωραία. Άρα μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. αποχε Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. αποχε Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ, 14 κατά. Συγγνώμη. 40 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 46 με προφορική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά Geschlossen. η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε 26 υπέρ καμία ψηφο, κατά, μία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μα. Πολύ ωραία θα ήταν να υπήρχε πάντοτε αυτή η συνένεση στην Επιτροπή μα. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Πολύ συχνά έχουμε εδώ συμφωνία μεταξύ μα. Τζούλι. My... Ναι, προηγουμένω σήκωσα το χέρι διότι δεν άκουγα την αγγλική μετάφραση, οπότε δεν άκουγα αυτά τα υπέροχα που έλεγες για μένα, Πέτρα. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στην πρώτη γραμμή και να κάνει ό,τι μπορεί για τα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών ε, διακυβεύονται και συρρυκνώνονται. Έγινε λοιπόν ε, πολύ καλή δουλειά, υπήρξε συνένεση και σας ευχαριστώ όλους. Ναι, και εγώ σε ευχαριστώ, Τζούλη, για τη δουλειά σου γύρω από αυτή την έκθεση πρωτοβουλία και ελπίζουμε τώρα η γνωμοδότησή μας να ληφθεί υπόψη από την ε, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Περνάμε λοιπόν στο θέμα 6, στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης. Όποιος θέλει να αποχωρήσει, παρακαλώ ας το κάνει αλλά ησύχως. Και θα μιλήσουμε τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα επόμενο ΠΔΠ, προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Η συγγήτριά μας είναι η Χέλγα Τρούπελ. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι η 17η Οκτωβρίου. 4 Δεκεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας. Επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Προεπολογισμού. Χέλγα, έχεις το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένα από τα βασικά, από τα καυτά ζητήματα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θα γίνει το 2020 όταν ε, πιθανότατα το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα έχει ε, αποχωρήσει. Μπορεί και να μείνει βέβαια, το εκτιμούσαμε αυτό, αλλά εάν φύγουν θα υπάρχει ένα κενό 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και δεν είναι σαφέ πώ θα το καλύψουμε. Έτσι λοιπόν οι επόμενε διαπραγματεύσει θα είναι ακόμα πιο σκληρέ από αυτέ ε, τη προηγούμενη δεκαετία και συμμετείχα σε εκείνε και μπορώ να σα πω ότι ήδη ήταν εξαιρετικά δύσκολε. Είναι δύσκολο να βρεθούν λύσει ε, με το Συμβούλιο. Τώρα, εμεί ω Επιτροπή είμαστε αρκετά ενωμένοι. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που ζητά περισσότερα χρήματα φρέσκο χρήμα για την εκπαίδευση, για την ε, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και έρχομαι τώρα στις συγκεκριμένες προτάσεις μου. Οι επόμενες διαπραγματεύσεις ε, θα λάβουν χώρα ε, σε ένα πλαίσιο χωρίς προηγούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά ένα από τα κράτη-μέλη αποχωρεί. Εφόσον δεν γίνει δεύτερο δημοψήφισμα, κάτι που δεν το ξέρουμε βέβαια. Αλλά εμείς πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα είμαστε χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Brexit λοιπόν αποτελεί πρόκληση για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων τη Ένωση. Ταυτόχρονα ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρία ε, έτσι ώστε να λάβουν χώρα οι μεταρρυθμίσει που χρειάζονται εδώ και πολύ καιρό στον προπολογισμό και σε επίπεδο εσόδων αλλά και σε επίπεδο εξόδων. Οπότε το θέμα είναι τελικά ε, πού δαπανούμε τα χρήματα και από πού προέρχονται. Είναι οι ίδιοι πόροι, παραδείγματο χάρη, μέσω ε, περιβαλλοντικών φόρων ή φόρων επί των συναλλαγών υπάρχει και έκθεση Μόντι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα παράθυρο, παράθυρο ευκαιρία για μεταρρυθμίσει. Ο κ. Ζώτη ήταν ανοιχτό προ αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια μικρή ελπίδα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Επίση η Ένωσή μα αντιμετωπίζει πολλαπλέ κρίσει τα τελευταία χρόνια που ζητούν νέε απαντήσει του ευρώ, της, την των νέων, της ασφάλειας, ε, το θέμα των προσφύγων και βεβαίως της αύξησης του λαϊκισμού. Ε, είναι κάτι που ε, κάνουμε, προσπαθούμε και εμείς να καταπολεμήσουμε την ε, ζωσβαστικοποίηση, να δώσουμε ευκαιρίες για τους νέους αλλά και για τους ενήλικους. Θα πρέπει λοιπόν με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση να προσεγγίσουμε τους πολίτες. Δεν πρόκειται να ερωτευτούν την ενιαία αγορά δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η Επιτροπή μα και νομίζω ότι το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Οι νέε αρμοδιότητε και, και πρωτοβουλίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ω αντίδραση στην κρίση πρέπει να αποτυπωθούν στις μελλοντικές... στο μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και αυτό είναι ένα θέμα που θα αποτελέσει ε, αντικείμενο συζήτηση ε, στι επόμενε ευρωεκλογέ, ε, είναι να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό project, να αποφύγουμε να επανέλθουμε στο κράτο έθνο. Ο εθνικισμό δεν είναι απάντηση στον 21ο αιώνα θα πρέπει τις κυριαρχίες μας να τις ενώσουμε δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις σε επίπεδο κράτους έθνους, ε, έθνους κράτους μάλλον ε, δεν είναι σωστή προσέγγιση αυτή. Πρέπει να πείσουμε του πολίτε, πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε για να γίνουμε μια καλύτερη και πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε βέβαια και τα μικρολικότητα, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ε, η εκπαίδευση, ο πολιτισμό, η ένταξη, πολύ σημαντικά στοιχεία. Είναι περιορισμένο το πεδίο βέβαια του σχεδίου γνωμοδότηση ε, ο στόχος όμως είναι να αρκετοκρίσουμε αυτό το πλαίσιο εντός των οποίων γράφονται οι πραγματεύσεις του, των, ε, ε, του πλαίσιου χρηματοδότησης. Ε, εκπαίδευση, παιδεία και έρευνα πρώτα. Εδώ έχουμε δύο βασικά επιχειρήματα. Οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δημοφιλία και προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το Erasmus Plus, χάρη, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ευρωπαϊκού προγράμματος και η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή λέγεται Σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης ε, ελπίζουμε ότι θα είναι άλλη μια εμβληματική επιτυχημένη πρωτοβουλία. Δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον λαϊκισμό, τον ε, εξτρεμισμό, τον ρατσισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, κοινωνίες ένταξης όσο γίνεται περισσότερο, όσο γίνεται πιο περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να απαντήσουμε καταλήλως ε, στην πρόκληση της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στις κοινωνίες μας, να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ε, ρόλο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης σε αυτό το ζήτημα. Αυτό πρέπει να, πρέπει να αποτυπώνεται ε, στο σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων για τον πολιτισμό. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να πείσουμε του συναδέλφου, να πείσουμε και το Συμβούλιο. που να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, αν θέλουμε να φτάσουμε κοντά στους πολίτε μα. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρο αυτού τη μελλοντική για τι ευρωεκλογέ του 2019. Τρίτον, πρέπει να ενισχύσουμε την ε, διάσταση από τους ανθρώπους προς τους ανθρώπους στον αφορά του Erasmus Αυτό ήδη το συζητούμε συχνά και τέταρτον θα πρέπει να εγκριθούν ε, έγκαιρα ε, τα πρόγραμμα και οι κανονισμοί για μετά το 2020 για να μην έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή των υπάρχουν προγραμμάτων. Ε, αυτό είναι θέμα ορθής διαχείρισης έτσι ώστε να αποφύγουμε τεχνοκρατικά, γραφειοκρατικά προβλήματα. Είναι θέμα απόδοση δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Χέλγα. Να προσθέσω και εγώ μια πληροφορία από τις συνεδριάσεις κλάστερ που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα με την Κομισιόν, όπου συνεδριάζουν οι πρόεδροι των Επιτροπών με τους, με τους μονομένους επιτρόπους και στη συνέχεια με το κολέγιο των επιτρόπων όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας της επόμενης χρονιάς κάθε φορά. Εγώ τουλάχιστον αποκόμισα την εικόνα ότι η Κομισιόν έχει κατανοήσει ότι πρέπει να υποβάλει τις προτάσεις για τα προγράμματα εντός του πρώτου τριμήνου του 2018. Είχαμε αποστείλει και μια σχετική επιστολή. Ε, νομίζω ότι αυτό έγινε κατανοητό. Εγώ ρώτησα προσωπικά και τον ε, Έτιγκερ και μου απάντησε ότι ναι, το καταλάβαμε, ότι προκειμένου να μπορείτε εσείς να ξεκινήσετε να, ε, το έργο σας, μπορούμε να σας στείλουμε τις προτάσεις για τα προγράμματα και χωρίς αριθμούς, χωρίς συγκεκριμένα νούμερα δηλαδή, για να μπορεί να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Και αυτό που επίσης έχει γίνει κατανοητό και εκεί όπου έχουμε μάλλον έναν σύμμαχο στην ε, Επιτροπή είναι η σημαντική αύξηση των κονδυλίων για το Erasmus+. Είναι ένα θέμα που τονίστηκε από πολλούς επιτρόπους στις ε, σχετικές συζητήσεις που είχαμε και φαντάζομαι και ελπίζω ότι τα λόγια δεν θα παραμείνουν λόγια αλλά θα γίνουν και πράξεις. Βεβαίως από εκεί και πέρα τα προβλήματά μας δεν έχουν τελειώσει. Θα πρέπει να πείσουμε και το Συμβούλιο ότι η επένδυση στο Erasmus Plus είναι μια ε, πραγματικά σημαντική επένδυση στο μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αυτά ε, όσον αφορά τις ε, συνεδριάσεις που έγιναν ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις συζήτητες. Ο κύριος Στρογεύσκη έχει το λόγο για δύο έως τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήταν ε, ε βεβαίως ε, πολύ εύκολο για μένα να συμφωνήσω με όλα αυτά που άκουσα ε, σε σχέση με αυτά που, που αναφέρονται στο έγγραφο όμως. Νομίζω πως είμαστε πολύ διστακτική στην ομοδότησή μα, Μιλάμε για πολύ κρίσιμα ζητήματα. Τι είναι το πιο σημαντικό για μα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε μια μάχη, μια ένα σταθερό προπολογισμό. Ένα σταθερό και ενισχυμένο προπολογισμό. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσει στι πληρωμέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν στο σημείο 1 πρέπει να ζητήσουμε έντονα το Erasmus Plus να διατηρηθεί όπως είπε και, ο, και η πρόεδρος, είναι, είναι ζωτική σημασία στο Erasmus Plus για την εικόνα της Ένωσης, για την ε, ε, φήμη της, ό,τι και αν γίνει λοιπόν, Brexit, εξοικονομήσεις, ε, περικοπές, το Erasmus Plus πρέπει να τα κομπήσει κανείς, δεν πρέπει να μειωθούν οι πόροι εκεί. Επίσης πρέπει να αναπτύξουμε την δημιουργική Ευρώπη. Το πρόγραμμα Creative Europe δεν είναι μόνο μια καλή πηγή για τα διάφορα ζητήματα που αναφέρονται στο σημείο 2 είναι μια ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε ότι ο πολιτισμός είναι ένας χώρος δημιουργίας είναι και μια οικονομική δραστηριότητα δηλαδή μπορεί να υπάρξουν και κέρδη από αυτόν τον τομέα από αυτόν τον κλάδο τρίτον μην ξεχνάμε ότι Έχουμε μια συζήτηση μπροστά μα για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να ζητήσουμε τα προγράμματά μας ε, να τοποθετηθούν κάπως καλύτερα, διότι συχνά στον προπολογισμό παραμελούνται. Θα πρέπει να απαιτήσουμε ε, να ανέβουν πιο, πολλά, πιο ψηλά προτεραιότητες. Τώρα, το θέμα της ευελιξίας. Συχνά λέγεται ότι τα προγράμματα στον τομέα του τουρισμού, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης ε, ότι τα προγράμματα αυτά είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν όπως το πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Κληρονομιά παραδείγματος χάρη και διαρκώς ε, υπάρχει μια τάση ε, να αποψηλώνονται τα προγράμματα αυτά. Τώρα με το Brexit θα πρέπει να τονίσουμε ότι όχι, όχι μόνο το Brexit δεν μπορεί να υπονομεύσει ε, τις οικονομικές πτυχές, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το Brexit δεν θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης όσων εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχουν ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο εργασιακό, διότι αυτό οδηγεί σε οικονομικό κόστος. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές τώρα, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, συχνά είναι το πιο επίπονο και το πιο δύσκολο ε, για τους δημιουργούς. Εδώ μιλάμε για μικρές οντότητες ε, που δεν μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν, πρέπει λοιπόν να μην υπάρχουν καθυστερήσει πληρωμέ. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι οι διαδικαστικέ ε, ε πτυχέ ε, θα αντιμετωπιστούν καταλήλω. Λουίτζι Μοργάνο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι μετά το 2020 μπορούν να γίνουν σημαντικές καινοτομίες ε, στην σύσταση του δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να επιμείνουμε για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το να δώσουμε, να παρέχουμε δημόσια ευρωπαϊκά αγαθά συμφωνεί με αυτά που είπε και η, η κυρία Τρούπελ, η συνάδελφος Τρούπελ, ενάντια στους ε, εθνικισμούς ενάντια ε, στους διχασμούς, να δείξει δηλαδή πραγματικά στους πολίτες τι είναι πραγματικά η Ευρώπη. Και έπειτα μία ερώτηση σε, συμφωνία με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην έκθεσή του για την κατάσταση της Ένωσης ότι θα πρέπει να είναι πολύ δημοκρατική η διαδικασία έγκρισης αλλά και να γίνεται και συγκεκριμένη αναφορά στην διάρκεια. Τώρα για τις προτεραιότητες βεβαίως Πάλι στα ίδια πράγματα επιμένουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η κινητικότητα έχει νόημα. Και άρα λοιπόν και αυτά οδηγούν και βοηθούν στο να οικοδομηθεί μια διαφορετική εικόνα για την Ευρώπη, ένα διαφορετικό όραμα. Αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στην έννοια της ηθαγένειας, στην αίσθηση της ηθαγένειας και για το θέμα της κινητικότητας πιστεύω συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα από αυτή την αντίληψη που επικρατεί σήμερα, ότι δηλαδή η κινητικότητα του εράσμου είναι βασικά μια κινητικότητα πανεπιστημιακή. Ενώ ήδη δεν συνισχύει αυτό, Υπάρχει θέμα κατανόησης, επικοινωνίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε ε, και να καταστήσουμε σαφές αυτό το στοιχείο. Επιμείνω όμως και για το εξής. Για να ε, ξεπεράσουμε τις ανισότητες και που είναι ένα θέμα που φυσικά και δικαίως βλέπει τους Ευρωπαίους πολίτες να αντιδρούν, θα πρέπει να τονίσουμε τον κοινωνικό πυλώνα που τον έχουμε ήδη εγκρίνει. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αν και είναι θέμα το με το οποίο ασχολούνται και άλλες επιτροπές. Αυτό σημαίνει ενίσχυση των προγραμμάτων για την εγγύηση για τους νέους και ιδιαίτερα το κονδύλι για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ενίσχυση του προγράμματος στήριξης για την πολιτιστική ε, παραγωγή. Ήδη αναφέρθηκε το θέμα της ε, δημιουργικής Ευρώπης, της Ευρώπης για τους πολίτες ε, και νομίζω πρέπει να επιμείνουμε και για το θέμα της δημιουργίας μιας εγγύησης για τους ανήλικους. Όλοι συμφωνούμε, όλοι λέμε πως είναι προτεραιότητα. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Το βαθύτερο πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι να, να επιτύχουμε να επιμείνουμε ώστε να βοηθήσουμε στην επίτευξη των γενικών στόχων επιμένοντας για παράδειγμα και στην Ε, στο πού θα δοθούν τα χρήματα στην, στον πολιτισμό. Το να περάσουμε από τον τίτλο 3 στον τίτλο 1 σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό νόημα. Κατανοώ ότι είναι ένα αίτημα αναγκαστικό, ότι δηλαδή όποιος κάνει προϋπολογισμούς ε, τα σκέφτεται διαφορετικά τα πράγματα. Επειδή όμω εμείς πολλές φορές έχουμε γκρινιάξει ότι ο πολιτισμός δεν αξιοποιείται, δεν έχει μπει στα σημεία που κανονικά θα έπρεπε να είναι, δηλαδή μέσα στις προτεραιότητες, κάποιοι είπαν επειδή είναι οριζόντιο ζήτημα. Ε, ζητάμε λοιπόν τότε μια απόδειξη ότι όντως ε, θεωρείται σημαντικός ο πολιτισμός. Να περάσουμε λοιπόν πρώτα από τους στόχους και την πρώτα από τους στόχους και μετά στον καθορισμό των κονδυλίων δεν γίνεται και με μηδενικό κόστος. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος Τόμ από τους φιλελεύθερους δεν είναι εδώ, ούτε η κυρία Νηριάντα. Κυρία Μπίλτ, θέλετε το λόγο? Euh, Μάλιστα, εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Συχνά είπαμε ότι έπρεπε να φτιάχνουμε πιο σαφή προγράμματα και δεν βλέπω καμιά αναφορά του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν αυτό να το βάλουμε χωριστά, να μην το προσθέσουμε τελευταία στιγμή όπως την τελευταία την περασμένη φορά. Και στην παράγραφο 4 υπάρχει μία φράση που λέει προτείνει μία αυτή για διαπροσωπική σχέση λοιπά. Δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτής της φράσης. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Η κυρία Σόντροβα έχει το λόγο για ένα με δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με την έκκληση του συναδέλφου και Πιστεύω πως το Brexit δεν μπορεί να είναι μόνο ένα αρνητικό στοιχείο μειώνονται τα χρήματα και οι άνθρωποι. Αλλά θα πρέπει επίσης να πούμε πως αυτές τις απώλειες θα πρέπει να τις ελαχιστοποιήσουμε ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν τα χρήματα και οι άνθρωποι και ότι τα όσα αντιπροσωπεύει η Μεγάλη Βρετανία για την Ευρώπη αυτή η απώλεια να ελαχιστοποιηθεί. Η συνάδελφος πολύ καλά είπε στην, στην τρίτο εδάφιο, λέει, για επενδύσεις. Εμείς ως, Ευρωπαϊκή, ως ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να τονίσουμε ότι το έρασμο ΣΥΝ είναι ε, θετικό και η Δημιουργική Ευρώπη επίσης γιατί σημαίνει επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε και θα πρέπει και τα κρατημέλη να το αντιληφθούν έτσι. Εάν θέλουμε να πείσουμε λοιπόν και εφόσον λέμε πως χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για αυτά τα προγράμματα, οφείλουμε να πούμε ότι κάνουμε επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο για τη βελτίωση της κατάρτισης, της προσβασιμότητας, της παιδείας, της, του πολιτισμού. Επενδύουμε στην ψηφιοποίηση του πολιτισμού. Είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και άρα λοιπόν θέλουμε να να δούμε αυτή τη λογική της αύξησης που ζητάμε μέσα στη λογική των, της επένδυσης. Η συνάδελφος ανέφερε την ε, μετανάστευση, τον αγώνα κατά της ε, κτλ. και τα λοιπά. Εκεί είναι ένας μόνιμος αγώνας. Η ψηφιοποίηση θα είναι όμως πολύ σημαντική για το μέλλον και χωρίς επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα στο μέλλον και πιστεύω πως αυτό το καταλαβαίνουν τα κρατημέλη. Ευχαριστώ πολύ. Σίλβια ένα με δύο λεπτά. Συμμερίζομαι τις απόψεις που τόνισε η συγγήτρια Τρούπελ, αν και πιστεύω πως θα πρέπει να αναφερθούμε με πιο έντονα κάποια πράγματα. Εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε κυρίως για κάποια πράγματα όπως το κάναμε στο ψήφισμα το πρόσφατο στην Ολομέλη για το θέμα του Εράσμους ένα έντονο μήνυμα ισχυρής συμμαχίας από πλευράς της Ευρώπης, συμμαχίας για τις νέες γενιές, για μια Ευρώπη που να είναι πιο ελκυστική και πιο φιλική στον πολίτη, να υπάρχει προσφορά ε, ποιοτικής ε, κατάρτισης και ε, δεξιο, ε, δεξιο, απόκτησης δεξιοτήτων, με συγχωρείτε. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε και να εστιάσουμε την προσοχή στην εφαρμογή του προϋπολογισμού αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περνά κρίση ταυτότητας ε, ώστε να παίξουμε πιο κεντρικό ρόλο. Γι' αυτό πιστεύω πως θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε η τόλμη να πούμε ότι όχι μόνο ε, ε θέλουμε να στηρίξουμε το έρασμος, αλλά θέλουμε να το πολλαπλασιάσουμε. Στο πέμπτο σενάριο, να θυμίσω, του λευκού βιβλίου του Γιούνκερ, που αναφέρεται και στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ε, μίλησε ότι θέλουμε να φτάσουμε στο 30% των νέων στην κινητικότητα το 2020. Σήμερα έχουμε μόνο το 5% και οι νέοι το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για πολλαπλασιασμό τουλάχιστον στην, στο ψήφισμα. Να έχουμε την τόλμη να ισχυριστούμε ότι εδώ υπάρχει όντως αλλαγή ε, ρυθμού. Το έρασμος δεν είναι περισσότερη παρουσία των ε, σχολείων, των πανεπιστημίων. Ξέρουμε πως υπάρχει εθελοντισμός, υπάρχει και αθλητισμός. Κάτι άλλο που θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να έχουμε εδώ ειδικό και συγκεκριμένο προϋπολογισμό και ε, το άλλο Δημιουργική Ευρώπη και προγράμματα για τον πολιτισμό. Και αυτό που είπε η και το, το συμμερίζουμε μετά από το ευρωπαϊκό έτος θα πρέπει να σκεφτούμε την προοπτική που θα έχουμε μετά το 2019 θα έχουμε τη νέα ατζέντα για τον πολιτισμό που θα πρέπει να λάβει υπόψη τους στόχους και τις στρατηγικές που έχουμε ε, ε, εγγενιάσει οριζόντια ε, θα πρέπει λοιπόν να το ξαναδεχτούμε. Είναι μια νέα προοπτική που έχουμε ανοίξει. Συμμερίζομαι αυτή την πρόταση κλείνω που φαίνεται να είναι κάπω προκλητική αλλά είναι πολύ σημαντική. Αυτή τη στιγμή η κουλτούρα είναι στο 3 και πρέπει πάντα να μοιράζεται με τη μετατενάστευση, την ηθαγένεια κτλ. Εγώ νομίζω πω θα ήταν ε, πολύ σημαντικό μήνυμα να πάει στην πρώτη, στον πρώτο τίτλο, δηλαδή επενδύσεις ανταγωνιστικότητα. Ίσως μπορούμε λοιπόν να δώσουμε αυτή τη μάχη μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Μέσιος. Μάθιος. Ως Βρετανός είμαι μεγάλος θαυμαστής του ευρωπαϊκού πολιτισμού και γι' αυτό χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σε αυτήν την Επιτροπή. Ωστόσο, ε, από τότε που έχω έρθει εδώ, ε, απογοητεύομαι πολύ από το γεγονός ότι διαπιστώνω ότι ε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ή πολλοί άνθρωποι εν πάση περιπτώσει δεν ε, μπορούν να αποδεχθούν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε μακριά. Θα είμαστε σύμμαχος και φίλος, αλλά δεν θα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί ως προς την ε, συζήτηση που γίνεται. Ε, ας μην φτιάχνουμε καρικατούρες, ε, σκιάχτρα με τα οποία αντιπαρατηθόμεθα, θέμεθα. Ε, γιατί νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε μόλις αποτελεί επιτομή αυτής της λογικής. Ε, της λογικής. Φυσικά και υπάρχει επικορικότητα, αλλά και μετά ε, ακούστηκε ε, ακούστηκαν διάφορα επιχειρήματα για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα κεντρικά. Μα άμα δεν κατανοήσετε ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα, θα το επαναλάβετε αλλού. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πραγματικά πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο Erasmus Plus, να ε, σκεφτούμε ε, καινοτόμους τρόπους για το οποίο, με τους οποίους μπορούν φοιτητές και ακαδημαϊκοί να συνεργαστούν διασυνοριακά. Ωστόσο, ε, αυτό, η απάντηση δεν είναι ε, απαραίτητα σε μια υπερεθνική οργάνωση ε, όπως αυτή την οποία εγκαταλείπει τώρα η Βρετανία. Η απάντηση βρίσκεται στις ψυχές των ανθρώπων, στα μυαλά των ανθρώπων και στην συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των κοινοτήτων των ανθρώπων και όχι απαραίτητα σε ένα τέτοιο μεγάλο κτίριο ή ένα μεγάλο θεσμό όπως αυτός εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάθιους. Ε, δεν είναι ότι δεν αποδεχόμαστε το γεγονός ότι αποχωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσα ίσα λυπούμαστε. Βεβαίως έχει και επιπτώσεις μια τέτοια απόφαση και η θέση του Κοινοβουλίου κατέστη σαφή στο ψήφισμα που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, και ε, όπου αναφέρεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να αναλάβει τις ευθύνε του για τις αποφάσεις του βεβαίως. Η θέση αυτή είναι σαφής, αυτό χωρίς, χωρίς καθόλου να σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε την απόφαση του, του Ηνωμένου Βασιλείου. Η απόφαση ελήφθη, πρέπει να το πάρουμε απόφαση όλοι μας. Κύριε Όφλιν. Um, Ευχαριστώ ε, κάποιοι ζουν στα σύννεφα νομίζουν ότι το Brexit θα μειώσει το επίπεδο χρηματοδότηση ε, στα πολιτιστικά προγράμματα. Ε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από του βασικού συνεισφορεί. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα έχει μια μαύρη τρύπα περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τα πολιτιστικά προγράμματα πρέπει να δεχθούν μέρος ε, της ε, των περικοπών. Ορισμένε φορέ βεβαίω μέσω τη μυρικότητα μπορούν να καλυφθούν κάποια από τα κενά. Αλλιώ ε, θα αυξηθούν ε, οι συνεισφορέ ε, των υπόλοιπων χωρών και αυτό δεν θα είναι βεβαίω αποδεκτό από τι εθνικέ κυβερνήσει. Και επίση θα μειώσει και την εικόνα τη Ένωση. Βλέπουμε ότι υπάρχει, λέμε εδώ, αύξηση τη ξενοφοβία, του εξτρεμισμού, του ρατσισμού αλλά η πλειοψηφία του εξτρεμισμού και της βίας προέρχεται από τους Ισλαμιστές που έχουν μεταναστεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται αναφορά ε, στα προβλήματα που προσφυγάζει η ένταξη για τους πρόσφυγες και τους ε, ε μετανάστες. Ε, ε, πρέπει αυτοί που έχουν αποφασίσει να έρθουν να ζήσουν εδώ να δεχτούν τις αξίες μας, τις πολιτιστικές. Ισότητα των δύο φύλων, ε, δημοκρατική πολιτική, ελευθερία έκφρασης. Οι λαοί της Ευρώπης ε, δεν είναι ότι ξαφνικά έγιναν κακοί ε, και είναι αρνητική απέναντι στους ξένους. Αυτό έχει να κάνει με μέρη και με τη συμπεριφορά των νέων, των νέων αφιχθέντων. Δεν πρέπει λοιπόν να αναπρογραμματίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για να σκέφτονται αυτά που είναι αποδεκτά πρέπει να ε, καταλάβουμε και να έρθουμε πιο κοντά στο πώς ε, ε, ζουν αυτοί οι άνθρωποι για να τους καταλάβουμε καλύτερα. Η κυρία Λιμπάτσκα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια αυτά που έχουν ήδη ελέγχθησαν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την δήλωση των Σαδέφων του Βασιλείου, ε, θα αλλάξω ριζικά αυτά που σκοπεύα να πω. Ε, είναι προφανές ότι η κάθε απόφαση οδηγεί σε κάποιες επιπτώσεις και δεχόμαστε και καταλαβαίνουμε την απόφαση των Βρετανών ή μέρος των Βρετανών εν πάση περιπτώσει αλλά ποτέ δεν πρόκειται να σκεφτώ ότι αυτοί που ψήφισαν υπέρ του Brexit ε, θέλουν ε, τα Βρετανικά πανεπιστήμια και οι Βρετανοί φοιτητέ να μην συμμετέχουν στον κοινό πανεπιστημιακό χώρο τον ευρωπαϊκό. Ε, δεν μπορώ με τίποτα να πιστέψω ότι αυτοί που ψήφισαν υπέρ του Brexit ψήφισαν να μην μπορούν οι Βρετανοί φοιτητέ να συμμετέχουν στο Erasmus Plus και στο πρόγραμμα κινητικότητας και ποτέ δεν πρόκειται να πιστέψω ότι όσοι ψήφισαν υπέρ του Brexit δεν θέλουν η βρετανική κουλτούρα, ο βρετανικός πολιτισμός να αποτελέσει μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Στα πλαίσια λοιπόν του Brexit και τη μείωση των πόρων αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα επηρεάσει και τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Θέλω να το πω για άλλη μια φορά, διότι δεν μπορώ πραγματικά να πιστέψω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να μην συμμετέχει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, αλλά μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ζωή δημιουργικά, συμμετέχοντας στον πολιτισμό και ε, στον, στην επιστημονική έρευνα. Η Σαμπίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συγκινούμε όταν βλέπω ε, πόσο ε, προβληματίζονται οι Βρετανοί συνάδελφοι για τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις αποχώρησής τους από το δημοσιονομικό πλαίσιο, από την Ένωση και οι επιπτώσεις για το ΠΔΠ. Πραγματικά με εξέπληξε ε, ο προβληματισμός αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας σοβαρευτούμε. Νομίζω ότι το θέμα δεν ήταν ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει κάποιες συγκεντρωτικές δομές για τον πολιτισμό. Αντίθετα, στόχο στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διατηρηθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία και πολυμορφία. Και γι' αυτόν τον λόγο ε, αξιοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει και αναπνέει και από την ανταλλαγή και την συνάντηση ανθρώπων, την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών, το να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον. Και αυτό ε, είναι και ένα στοιχείο που μπορούν να το επιβεβαιώσουν ε, και οι ίδιοι οι Βρετανοί πρώτοι από όλου, καθώς και οι ίδιοι έχουν έρθει σε επαφή ιστορικά με πάρα πολλούς λαούς ε, στους οποίους, στον πλανήτη στους οποίους, ε, με τους οποίους ε, είχαν πολύ στενές σχέσεις. Αυτό βεβαίως ε, δεν αναιρεί το γεγονός ότι εμείς ε, έχουμε υποχρέωση να καταρτήσουμε το μελλοντικό μας προϋπολογισμό και χωρίς τη Βρετανία και ε, όταν πια ξεκαθαριστούν οι όροι της αποχώρησης θα προχωρήσουμε και ως προς το θέμα των μελλοντικών δομών συνεργασίας και εδώ υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για την ενισχυμένη συνεργασία και επαφή μεταξύ φοιτητών, πολιτών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν ε, μια συνεργασία επί δεκαετίες και το γεγονός ότι εμείς θέτουμε αυτά τα θέματα στο επίκεντρο νομίζω ότι είναι σαφές και δικαίωμά μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε άλλους δύο-τρεις ε, ομιλητές. Και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή γιατί στις 10 έχουμε ε, προσκαλέσει μια, ε, ε, έχουμε προσκεκλημένη ε, την οποία και δεν θα ήταν σωστό να καθυστερήσουμε. Julie Ward. Εγώ είμαι υπερήφανη Βρετανίδα και Ευρωπαία και ντρέπομαι που υπάρχουν στην αίθουσα αυτή άνθρωποι που υποβιβάζουν και υποβαθμίζουν τόσο πολύ το ευρωπαϊκό εγχείρημα που αφορά την ειρήνη και την αρμονία. Εγώ δεν, έχω, δεν προέρχομαι από τον ε, κομματικό σωλήνα. Αντιθέτως ε, έχω εργαστεί και δραστηριοποιηθεί στη Βόρεια Αγγλία, στη βάση ε, και γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πολιτιστικά προγράμματά της που προσφέρθηκαν σε νέους ανθρώπους, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά σε ολόκληρη την Ήπειρο, ε, έχουν αποτελέσει μια πολύ δυνατή εμπειρία. Έχουν βοηθήσει νέους ανθρώπους να ε, έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Διότι όταν μαθαίνεις για τον άλλον, μαθαίνεις πολλά πράγματα για τον, αυτές, για τον αυτό σου. Το γεγονός λοιπόν ότι το ε, Brexit, η καταστροφή αυτή που ε, ε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως είδαμε και στο συνέδριο των συντηρητικών την προηγούμενη εβδομάδα. Η Τερέζα Μέη μάλιστα έχει περιγράψει το Brexit ως κάποιο ομαδικό άθλημα με μπάλα. Ε, βρισκόμαστε ε, λοιπόν σε μεγάλους μπελάδες, Βρετανοί συνάδελφοι, σε εσάς απευθύνομαι. Δεν είναι λοιπόν η δική μας γενιά, ούτε εσείς αυτοί που θα κληθούμε να πληρώσουμε το αντίτιμο. Είναι οι νέοι άνθρωποι και πραγματικά ε, ε, ντρέπομαι που βρίσκεται σε αυτή την επιτροπή ο Πάτρικ Όφλιν με τις ισλαμοφοβικές του απόψεις με τις ομοφοβικές του απόψεις και εγώ ε, χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ε, επισκέπτρια εδώ μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, μια νέα κοπέλα την οποία και σας καλώ να συναντήσετε και να της τα πείτε κατά πρόσωπο, διότι είναι πραγματικά ντροπή να έρχεστε και να λέτε εδώ στο Κοινοβούλιο αυτά τα πράγματα, αυτές τις απόψεις. Ευχαριστώ, ο κύριος Διακονού έχει το λόγο. Υπάρχει μια σημαντική ερώτηση. Τι είναι ένας εγωιστής άνθρωπος. Αυτό είναι, η απάντηση είναι, είναι αυτός που φροντίζει περισσότερο τους άλλους παρά τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι κάτι το αντίστροφο, αλλά ένα πολιτιστικό ζήτημα ε, μετατρέπεται σε ένα τελείως βρετανικό ζήτημα εδώ η Βρετανία αποφάσισε και είμαστε βέβαιοι πως θα τα καταφέρουμε και από εδώ και μπρος όπως κάναμε άλλωστε μέχρι τώρα. Θυμάμαι ως ε, επιχείρημα με τις διαπραγματεύσεις με τους υπολείπους ότι η, τα μεγάλα οικονομικά άλματα βασίζονταν σε απλά πολιτιστικές, πολιτιστικά νοη, ε, κινήματα, δηλαδή αναγέννηση, διαφωτισμός, ήταν πολιτιστικά κινήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, προγραμμάτιζα να παρέμβω, αλλά αφού άκουσα όλο αυτό το βρετανικό πάθος για λίγο, πιστεύω πως ε, ένα σύντομο προβληματισμός θα ήταν σωστός. Να θυμίσω σε όλους ότι θα δούμε αύριο μεθαύριο, μετά το Brexit, τι θα γίνει. Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το δεύτερο μεγαλύτερη σημαντική χώρα στο ΝΑΤΟ, τεράστια επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο, θα πνιγεί στον Ατλαντικό. Φυσικά και όχι κέρδισε δύο παγκόσμιους πολέμους ε, και έβαλε τα γελιά στον Ναπολέοντα. Και μετά τον Brexit λοιπόν η Βρετανία θα σταθεί οικονομικός, πολιτικός ε, και θα φωτίζει τον κόσμο ω φάρο. Και δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί σε αυτόν τον ενθουσιασμό σα, ε, για αυτό το καταπληκτικό σα ευρωπαϊκό project, αυτό ο φωτεινό φάρο μπορεί να αποτελέσει καλύτερη εναλλακτική, όχι σήμερα, όχι σε ένα χρόνο, αλλά σε 5-6 χρόνια να αποτελέσει καλύτερη εναλλακτική για άλλα μέλη αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν ακούσετε ή αν δεν βελτιωθείτε. Και η μόνη σας υπεράσπιση για αυτό που έχετε σήμερα είναι να κουνάτε τα σκιάχτρα και να λέτε ότι είμαστε ισλαμοφοβικοί ε, και καημένοι, τότε είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από ό,τι φανταζόμουν πριν να έρθω στη σημερινή αυτή συνεδρίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά κανείς εδώ στο Κοινοβούλιο ε, δεν τηρεί μια στάση μη σεβασμού προς την αποχώρηση της Βρετανίας. Το αποφάσισε ο Βρετανικός λαός. Λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό που έχουμε εμείς ως καθήκον να κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διαμορφώσουμε τους όρους αυτού του διαζυγίου. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Όταν ολοκληρωθούν θα έχουμε να συζητήσουμε ε, ποια θα είναι η μελλοντική μας σχέση με τη Βρετανία. Και δεν ε, άκουσα κανέναν να προσπαθεί να υποβαθμίσει, να υποβιβάσει ε, την αξία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντιθέτως, είπαμε ότι σεβόμαστε την απόφαση, ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε ε, σε πνεύμα αμοιβαίου ωφέλους το τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση αυτού του διαζυγίου. Και γι' αυτό θέλω να ξανατονίσω αυτό που είπε η Ζαμπίνε Φερχάιεν, το ότι είναι πραγματικά ε, εντυπωσιακό το πόσο συμμετέχουν οι Βρετανοί ε, συνάδελφοι σε όλες τις συζητήσεις που αφορούν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το επόμενο. Δεν θα είστε πλέον εδώ. Αφήστε μας λοιπόν και εμάς να συζητήσουμε το θέμα αυτό και άπαξ και αποχωρήσετε οριστικά πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε όλο το χρόνο και όλες τις δυνατότητες να ε, διαμορφώσουμε την μελλοντική μας σχέση. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην Κομισιόν και στο τέλος ξανά στην Χέλιγκα Τρούπελ. Εγώ δυστυχώς πρέπει να ε, φύγω για 15 λεπτά θα επανέλθω όμως ε, και ευχαριστώ πολύ την Χέλγα Τρίπελ που δέχτηκε να αναλάβει την ε, Προεδρία της ε, Επιτροπής για το μικρό αυτοχρονικό διάστημα. So Λοιπόν, τον λόγο έχει η Κομισιόν. Παρακαλώ. Je vous remercie de donner Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αν μου το επιτρέπετε, πολύ σύντομα θα μιλήσω Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης εξαιρετικά σημαντικό. Θα συνεισφέρει ελπίζω να επερασπιστούμε τη θέση των προγραμμάτων μας στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μεταξύ των μελλοντικών προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού της Ένωσης μετά το 2020. Παρακολουθούμε τη συζήτησή σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως αντιλαμβάνεστε. Επίσης ε, ακούσαμε τις προτάσεις ε, δημοσιονομικής ενίσχυσης. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για την συνεισφορά της, η οποία είναι θεμελιώδης, έτσι ώστε να αυξηθεί όσο γίνεται περισσότερο ο αντίκτυπος του Erasmus Plus και του Creative Europe, καθώς και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ε, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τώρα το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 13 Σεπτεμβρίου, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για το μελλοντικό πλαίσιο που προβλέπει ότι η Κομισιόν θα υποβάλει την πρότασή της ε, το Μάιο του 2018. Παράλληλα θα γίνει μια σημαντική συζήτηση επί του συνόλου των προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών μέσων ε, που προέρχονται από τον προπολογισμό της Ένωσης μια συζήτηση που θα οδηγήσει συμπεράσματα στο δεύτερο εξάμεινο του χρόνου όταν η Κομισιόν θα υποβάλει συγκεκριμένε προτάσεις ιδιαίτερα για το Erasmus Plus την Creative Europe αλλά και το Σώμα Αλληλεγγύης. Εν τω μεταξύ βεβαίω θα χρειαστεί χρόνος έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας ε, τα διδάγματα από την εφαρμογή των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της παρούσας, ε, της τρέχουσας περίοδου αλλά και των δημοσιονομικών επιπτώσεων του Brexit αλλά και της εισαγωγή ε, νέων προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δύο ζητήματα που συνδέονται μεταξύ τους υπάρχει μια άλλη λεξάρτηση. Τελειώνοντας να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να απλοποιήσει τα πράγματα, να είναι πιο αποτελεσματική στην εκτέλεση των προγραμμάτων, να υπάρχουν μεγαλύτερε συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων, να είναι πιο εύκολη προσβασιμότητα, να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο του κάθε ευρώ που ξοδεύουμε για τους πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να απλοποιήσουμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ξαναπέρνω το λόγο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, διότι πραγματικά ήταν μια πολιτική συζήτηση και σπάνια συμβαίνει αυτό στην Επιτροπή Πολιτισμού, περισσότερο στην Ολομέλεια. Ήταν χρήσιμο πάντως. Οι συνάδελφοι Μάθιους του EFFD, η κυρία Μπίλντε, θα ήθελα να κρατήσω σαφές, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, απευθύνομαι σε αυτούς, αποδέχομαι 100% το δημοκρατική επιλογή των Βρετανών πολιτών. 100% είναι δημοκρατικό δικαίωμά σα. Αν θέλετε να φύγετε, φεύγετε. Δεν μπορείτε όμω να είστε και μέσα και έξω ταυτόχρονα. Πρέπει να αναλάβετε και τι ευθύνε σα. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν μειονεκτήματα για του Ευρωπαίου πολίτε και του Βρετανού πολίτε. Εάν θέλετε όμω να φύγετε, φεύγετε. Σε πολιτικό επίπεδο βεβαίω εγώ λυπάμαι. Διότι θεωρώ ότι θα υπάρξουν πολλά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα για του Βρετανού πολίτε. Εσεί δεν συμφωνείτε. Εντάξει. Και αυτό το δέχομαι. Δέχομαι διαφορετική άποψη. Είμαι δημοκράτησα. Αλλά μπορώ να σας πω και εγώ ποια είναι η άποψή μου. Φύγετε και τις επιπτώσεις θα τις επομιστείτε. Αυτό είναι σαφές. Σε μερικά χρόνια, σε μια δεκαετία θα δούμε ποιος είχε δίκιο και ποιος όχι. Δεν είναι θέμα να μην δέχεται κάποιο μόνο δημοκρατικές δημοκρατικέ ψηφοφορίε. Τι δέχομαι πάντα τα, τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπω δέχομαι και τι αποφάσει των ε, Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, ακόμα και αν δεν μου αρέσουν. Διότι το κράτο δικαίου είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το πολιτικό ζήτημα. Κατά πόσο υπάρχει μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο μπορούμε να συνδέσουμε, να συνδυάσουμε ε, την υπερεθνική και την εθνική δημοκρατία, να έχουμε ταυτόχρονα και επικουρικότητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται, αλλά θα πρέπει όμω να έχουμε του πολίτε μαζί μα να αντιληφθούν ότι τον 21ο αιώνα δεν έχει νόημα να επιστρέψουμε, να στα εθνικά κράτη και στον εθνικισμό. Εσείς συμφωνείτε, το δέχομαι και αυτό. Η πολιτική μου προσέγγιση είναι να συνδυάσουμε το υπερεθνικό, το εθνικό επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο δημοκρατίας, το τοπικό επίπεδο δημοκρατίας και την επικουρικότητα. Αυτή είναι η διακυβέρνηση, η πολυεπίπεδη και αυτή χρειαζόμαστε 21ο αιώνα. Είμαστε λοιπόν σε μια διαφορετική, σε διαφορετικό μήκο κύματο. Το θέμα τη βία τώρα. Είναι πολύ πιο δύσκολο τα πράγματα από ό,τι λέτε. Δεν είναι μόνο η ριζοσπαστικοποιημένοι μουσουλμανοί. Υπάρχει πρόβλημα εκεί, αλλά υπάρχουν και αντισημιτε. Υπάρχει βία από ακροδεξιού, από ακροαριστερού και πρέπει όλου μα να του αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι δημοκρατικά πράγματα αυτά που θέλουμε να πετύχουμε εμεί τα προγράμματά μα με, τον, με την απορρασπιστικοποίηση είναι να αντιμετωπίσουμε όλε τι μορφέ βία ε, από τη δεξιά, από την αριστερά. Έχουμε την NSU ε, στο, στη Γερμανία. Είχαμε και τη ΡΑΦ στο παρελθόν, άλλε τρομοκρατικέ οργανώσει, ε, ακροαριστερέ, ακροδεξιέ, θρησκευτικέ, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν μπορέσουμε να τι αντιμετωπίσουμε, θα είναι καταστροφική κατάσταση και θα είναι επικίνδυνο για όλου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να δράσουμε επ' αυτού. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, στα πλαίσια τη εκπαίδευση του πολιτισμού και τη κοινωνική ένταξη. Και θέλω επίση να καταστήσω σαφέ ότι βεβαίως και μπορείτε να φύγετε, αλλά πρέπει να αποδεχθείτε τις συνέπειες. Και θα δούμε στη συνέχεια ποιος είχε δίκιο. Δεν είναι κάτι που θα αποφασιστεί όμως τώρα. Θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Και βεβαίως εγώ δεν αμφισβητώ το μεγαλείο του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας Είναι μια μεγάλη χώρα με καταπληκτική παράδοση είναι ένα ε, σημαντικό οικονομικό παίκτη, έχει τα προβλήματά του όπως και άλλα κράτη-μέλη, όπως το δικό μου κράτος μέλος, η Γερμανία. Και τώρα έρχομαι στου άλλους συναδέλφου ε, που δεν αφισβητούν ε, την ύπαρξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν να τη βελτιώσουν καθώ και τα προγράμματά μας. Έχετε δίκιο κύριε Σντρουγεύσκη, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, να μην είμαστε ε, άτολμη. Αναμένω λοιπόν τι τροπολογίε, σα Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη τόλμη και πρέπει να ανισχυθεί το Erasmus Plus, το Creative Europe και όλα τα λοιπά προγράμματα. Ε, θέλουμε ε, όντως ε, να υπάρξει μια δημόσια προσέγγιση και επίση έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, η ηθαγένεια, η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, όχι μόνο η εθνική, η εθνικιστική προσέγγιση και τα στήματα αυτά. Θέλουμε να έχουμε περισσότερες επαφέ από του ανθρώπου προς τους ανθρώπους, δηλαδή τους ανθρώπων μεταξύ τους, από κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω. Εγώ είμαι φιλελεύθερη, πράσινη, ε, θα μιλούσα περισσότερο για την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά εν πάση δεν έχει τόσο σημασία η διατύπωση ε, πρέπει να να σαφέ ότι η απασχολησιμότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, αλλά δεν είναι ο μόνο σκοπό όταν μιλάμε για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, διότι υπάρχει και μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την, ανθρώπινη, την ανάπτυξη κάποιων ανθρωπίνων δεξιοτήτων, που είναι πολύ σημαντικό να ε, ε, τονίσουμε. Θα συνεργαστώ μαζί σας σε αυτό το πνεύμα. Ε, ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Ωραία, περνάμε στο επόμενο θέμα. Θα μιλήσω στα γερμανικά γιατί το έχω προετοιμάσει στα γερμανικά. Α, έρχεται. Ωραία. Σημείο 7. Λοιπόν, ανταλλαγή με την ε, νέα Μέα Κίλοαν, ε, διευθύντρια του Κέντρου Μετάφρασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεια σας. Το επόμενο θέμα λοιπόν έλεγα ότι είναι ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Μέρ Κίλωραν, Διευθύντρια του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είναι αρμόδια και για ζητήματα πολυγλωσσίας. Ως προς αυτό το καθήκον μας λοιπόν, μας ενδιαφέρει πολύ το έργο του Μεταφραστικού Κέντρου. Στην τελευταία ε, συνεδρίαση των συντονιστών λάβαμε την απόφαση να ενισχύσουμε τις επαφές μας με αυτό το μεταφραστικό κέντρο. Επίσης, ε, εγκρίναμε μια γνωμοδότηση, ε, μάλλον ε, εγκρίναμε την σύνταξη μιας γνωμοδότησης για την απαλλαγή για το 2016. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κίλωραν για να μας ενημερώσει για το έργο του μεταφραστικού κέντρου. Έχετε 10 με 15 λεπτά περίπου, κυρία Κίλωραν. Παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για την ευκαιρία που μου δώσατε να, έρχομαι, να παρίσταμε εδώ στην συνεδρία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το έργο μας και ε, προφανώς και λόγω της πολυγλωσσίας που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει καλύτερο περιβάλλον από, από το δικό σας. Να σας ε, παρουσιάσω λοιπόν ε, το εύρος των δραστηριοτήτων μας, των, τους πελάτες μας και βεβαίως εν ώψη, και την, εν της ε, γνωμοδότησης που θα συντάξετε για την απαλλαγή για το 2016. Λοιπόν, δημιουργηθήκαμε το 1994 στο Λουξεμβούργο προκειμένου να παρέχουμε μεταφραστικές υπηρεσίες σε 7 πελάτες και ε, κατέστημεν επιχειρησιακή το 1995. Αργότερα, με τροποποιητικό κανονισμό το 1995, διευρύναμε τις δραστηριότητες μας προκειμένου να μπορέσουμε να ε, παρέχουμε αυτόνομες μεταφραστικές υπηρεσίες σε εθελοντική βάση με σκοπό να απορροφήσουμε ε, τυχόν περίσσια έργου από τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με επιπλέον εντολή να συμβάλλουμε στην θεσμική ε, συνεργασία. Πρόκειται λοιπόν για τον ε, κατεξοχήν πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. De facto λαμβάνουμε πληρωμές από οργανισμούς και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες μας. Δεν λαμβάνουμε συμβολή από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αν και κάτι τέτοιο προβλέπεται ε, ε, θεσμικά. Α, λοιπόν, έχουμε διοικητικό συμβόλιο, εγώ είμαι διευθύντρια και προφανώς λογοδοτώ σε αυτό το ε, συμβούλιο. Έχουμε διτό στόχο. Πρώτον, ως γλωσσικός πάροχος παρέχουμε μεταφραστικέ υπηρεσίε στου ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωση όσον αφορά την περίσσια έργου, που ε, ορισμένες φορές υπάρχει και ε, επίσης έχουμε ρόλο στην διοργανική συνεργασία και το συντονισμό. Ως ε, κοινός μεταφραστικός πάροχος δημιουργηθήκαμε προκειμένου να επιτύχουμε εξοικονομήσεις και να μην δημιουργούνται μικρές μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλους τους οργανισμούς. Ε, θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία και για την εξέλιξη του οργανισμού μας από τότε που κατέστημε ε, επιχειρησιακή το 1995. Η εξέλιξη λοιπόν αυτού του κέντρου ε, χαρακτηρίστηκε από την πολύ μεγάλη αύξηση του έργου της καθώς αυξήθηκε και μια, αυξήθηκε και πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό ο αριθμός των επίσημων γλωσσών. Φαίνεται εδώ σε αυτό το γράφημα ότι οι μεταφραστικές υπηρεσίες ε, βρίσκονται σε ευθεία συνάρτηση με τον, την αύξηση του, του αριθμού των επισήμων γλωσσών. Ε, από το 1995 λοιπόν έχουν αυξηθεί οι επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Να πω όμως ότι από το 2009 υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση του προσωπικού. Όπως γνωρίζετε η Δημοσιονομική Αρχή έχει επιβάλει 5% μείωση προσωπικού σε όλους τους οργανισμούς και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον η Κομισιόν έβαλε άλλο, άλλο έναν στόχο μείωσης 5% για τις νέες προσλήψεις. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν, έχουμε λοιπόν πολύ λιγότερο προσωπικό από ό,τι το 2009. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν την περίοδο 2012-2017 έχουμε 20 ε, θέσεις λιγότερες, 9,3% και μας ζητείται από την Κομισιόν να κάνουμε περαιτέρω μειώσει του προσωπικού. Αν ε, ληφθεί σχετική απόφαση από τη Δημοσιονομική Αρχή βεβαίως θα την ε, εφαρμόσουμε όπως και στο παρελθόν, ωστόσο ε, πρέπει να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, ίσα ίσα που καταφέρνουμε δηλαδή να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Κάθε περαιτέρω περιορισμός του προσωπικού θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας. Ποιοι είναι οι πελάτες μας. Έχουμε 65 πελάτες αυτή τη στιγμή, είναι οι οργανισμοί, θεσμικά όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με βάση τον ε, καταστατικό κανονισμό, ε, οι οργανισμοί αυτοί, όλοι αυτοί οι φορείς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούν να απευθύνονται στην, στον, στο μεταφραστικό κέντρο προκειμένου να εξυπηρετούνται, να καλύπτονται οι μεταφραστικές τους ανάγκες και καλύπτουμε όλους τους τομείς. Όσον αφορά τις υπηρεσίε, υπάρχει μια πλειάδα. Προφανώς είναι η μετάφραση, υπάρχει όμως και ο υποτιτλισμός και η συμβουλευτική όσον αφορά την ε, πολυγλωσία. Είναι σημαντικό να σας παρουσιάσω και το επιχειρηματικό μας μοντέλο, ε, διότι μας ενδιαφέρουν πολύ εξοικονομήσεις ε, χρημάτων. Όπως είπα, δεν λαμβάνουμε χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό μας μοντέλο, λοιπόν, είναι πολύ αποτελεσματικό, διότι οι περισσότερες μεταφράσεις μας ανατίθενται σε εξωτερικούς μεταφραστικούς παρόχους και στη συνέχεια η ποιότητα ελέγχεται από τους εσωτερικούς μας μεταφραστές προτού διαβιβαστούν προτού ε, αποσταλούν μεταφράσεις στους τελικούς ε, πελάτες μας. Επίσης, ε, σεβόμαστε πλήρως την πολύγλωση πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι γλώσσες για εμάς είναι ισότιμες. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος του outsourcing και μεταφράζουμε προς όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες αλλά και γλώσσες που δεν είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως βλέπετε σε αιτήσια βάζη μεταφράζουμε περίπου 750.000 σελίδες. Τεράστιο κομμάτι αυτών, αυτών των μεταφράσεων αφορά την, τον EUIPO, το το, τον Οργανισμό ε, Ευρεσιτεχνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότερες γλώσσες πήγε, ε, οι περισσότερα, τα περισσότερα κύματα ε, καταφτάνουν σε εμά στις πέντε μεγάλες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και από εκεί ε, μεταφράζονται σε όλες τις άλλες γλώσσες. Όσον αφορά το μοντέλο εξασφάλισης ποιότητας είναι πολύ αυστηρό. Ε, αυτό αφορά και τις προκηρύξεις ε, και εξασφαλίζουμε πάντοτε ότι έχουμε προσκλήσεις ε, εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους οποίους θα, στις οποίες θα συμμετέχουν μεταφραστικοί πάροχοι οι οποίοι θα μπορούν να, να παρέχουν και εξειδικευμένε επίρρησεις νομικές μεταφράσεις, τεχνικές μεταφράσεις και βεβαίως έχουμε και ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης ποιότητας αυτών των εξωτερικών συνεργατών. Ε, για το 2016, από τον Ιανουάριο του 2016 που ορίστηκα εγώ διευθύντρια, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε μία ε, πενταετή στρατηγική, ε, της οποίας όραμα είναι να ε, γίνουμε ένα κέντρο αριστείας όσον αφορά τη μετάφραση ε, για τους φορείς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2020. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι το 2016 αναπτύξαμε ένα νέο σύστημα ροής εργασιών, διαχείρισης των εργασιών, το οποίο ε, έχει τίτλο ECDT το οποίο, και το οποίο περιλαμβάνει ένα πορτφόλιο, ένα χαρτοφυλάκιο για τους πελάτες, ένα ε, χαρτοφυλάκιο για τους εξωτερικούς ελεύθερους συνεργατές μεταφραστές και ένα χαρτοφυλάκιο που αφορά την ροή και τη διαχείριση των εργασιών εσωτερικά. Όσον αφορά τον όγκο των μεταφράσεων του 2016 βλέπετε ότι περίπου 750.000 σελίδες μεταφράστηκαν τα εμπορικά σήματα αφορούσαν περίπου το 61% ενώ τα έγγραφα 38% του συνολικού έγκου των ε, εργασιών μας. Όσον αφορά τους πελάτες μας, ο μεγαλύτερος πελάτης που έχουμε είναι ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, για τη Διανοητική Ιδιοκτησία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός σερμάκων, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου. Θα ήθελα επίσης να σας δώσω κάποια στοιχεία όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας για το 2016, για να γνωρίζετε πού βρισκόμαστε και χρηματοδοτικά. Το 2016 ε, τα έσοδά μας ε, ήταν μεγαλύτερα από, τα, από, τα, τις δαπάνες μας. Ε, θέλουμε να, ωστόσο να δημιουργήσουμε ένα έλλειμμα, διότι συσσωρεύσαμε τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο ε, περίσσευμα στον προϋπολογισμό μας. Πώς το κάναμε αυτό. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε σταθερές τις μας, στις, τιμές μας, για να απαντήσουμε ε, στις μεγάλες διακυμάνσεις που εμφανίστηκαν στην αγορά της μετάφρασης. Ε, αποφασίστηκε λοιπόν να, ε, ε, από το 2015 να υιοθετήσουμε μια αρνητική ε, προσέγγιση ως προς το, προς το ισοζύγιο του προϋπολογισμού μας. Στην ίδια περίοδο η τιμή της, ε, του, που χρεώνουμε για την ανασελίδα ε, διακυμάνθηκε. Ε, βλέπετε εδώ στον ε, κανονισμό, ότι υπάρχει, στο, στη διαφάνεια αυτή, ότι υπάρχει και μια ευθεία συσχέτιση ανάμεσα στην τιμή που χρεώνουμε και ε, στα αποτελέσματα που είχαμε στα τέλη του κάθε έτους όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε και αυτό το περίσσευμα στον προϋπολογισμό μας τα τελευταία χρόνια το οποίο προσπαθούμε τώρα να ε, μετακυλήσουμε με τη μορφή καλύτερων τεμών ανασελίδα στους πελάτες μας. Οι, μας, οι τελευταίες μας εμπειρίες το τελευταίο 9 δηλαδή, μας δείχνουν ότι υπάρχει ε, μια, ένα σημαντικό, μια σημαντική μείωση του κόστους για τους πελάτες μας, ανασελίδα μετάφρασης, κάτι που βεβαίως τους χαροποιεί, χαροποιεί ιδιαιτέρως. Αυτό βεβαίως ε, σημαίνει ότι το, στο μέλλον, κατά πάσα πιθανότητα, η, η τιμή μετάφρασης ανασελίδα θα ξανααυξηθεί ε, διότι το πλεόνασμα του προπολογισμού δεν θα διατηρηθεί στο διηνεκές, άρα ε, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα αυξήσουμε την τιμή μας. Επίσης, όσον αφορά την πολυγλωσία, θα ήθελα να επισημάνω την ιδιαίτερη συμβολή του κέντρου μας στην πολυγλωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η πολυγλωσία είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά την ίδια της δημοκρατική νομιμοποίηση, την επικοινωνία της με τους πολίτες και το κέντρο μας διευκολύνει ακριβώς αυτήν την, την αποτελεσματική εφαρμογή της πολυγλωσσίας. Για παράδειγμα, η ε, βάση δεδομένων ΙΑΤΕ είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων ε, ορολογίας στον κόσμο. Ε, βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ε, ότι ε, οι αναζητήσεις που γίνονται ε, στο ΙΑΤΕ είναι τεράστιος ο αριθμός των αναζητήσεων που έγιναν. Ε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ε, φάση ε, δημιουργίας του ΙΑΤΕ 2 που θα διατεθεί στο κοινό το 2018. Πρόκειται για μια μορφή διοργανικής συνεργασίας που πραγματικά ωφελεί τους πολίτες. Όσον αφορά την, την ορολογία και τα, οπτικοαισθη την, την ορολογία βλέπετε εδώ ότι ε, ο ε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών ε, έχει δημιουργήσει πλέον μια βάση δεδομένων με τη βοήθειά μας η οποία είναι δημόσια προσβάσιμη και όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει όρους χημίας. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με ένα γλωσσάρι που αφορά την, την ισότητα των δύο φύλων. Και τέλος να σας αναφέρω το, την ε, εφαρμογή για κινητές ε, συσκευές της ΕΑΣΟ ε, που επιτρέπει σε ετούντες άσυλο να αναζητήσουν πληροφορίες στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου καλύπτονται πολλές γλώσσες πλήν των αγγλικών και τα αραβικά και άλλες γλώσσες. Αυτά. Όσον αφορά την σχέση μας με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έχουμε από το 2016 εκπονήσει διάφορες μελέτες για να δούμε ποια είναι η στάση των επιμέρους οργανισμών όσον αφορά την πολυγλωσία. Βλέπουμε ότι έχουν σημειωθεί κάποιες αλλαγές όσον αφορά τις πρακτικές που ακολουθούν διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί στον τομέα της πολυγλωσίας αλλά και στις ιστοσελίδες που συντηρούν οι οργανισμοί αυτοί. Και να αναφέρω στο τέλος επίσης και τη δική μας ε, ιστοσελίδα που βεβαίως ε, παρέχεται και στις 24 ε, επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν να σας έδωσα μια καλή εικόνα για το πού βρισκόμαστε και το τι κάνουμε και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Το μικρόφωνο της Προέδρου είναι κλειστό. Sorry. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση του έργου σας που ε, νομίζω ότι δεν είναι σε όλους ε, ιδιαίτερα γνωστή και από αυτή την άποψη ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η παρουσία σας και η παρουσίασή σας αυτή. Να δώσω το λόγο στον κύριο Στρογεύσκη που είναι ο εισηγητής μας για την απαλλαγή ε, του Κέντρου Μετάφρασης και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο και σε όλα τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας που θα τον ζητήσουν. Κύριε Στρογεύσκη, για δύο έως τρία λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Κιλοράν για αυτές τις πληροφορίες που μας ε, παρουσιάσατε. Φαίνεται ότι ήταν ε, καλή ε, απόφαση να εξαιρεθεί ο δικός σας οργανισμός από την ε, γενική έκθεση που συντάξαμε και το κάναμε αυτό ακριβώς για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις δραστηριότητές σας και τις αρμοδιότητές σας. Δεν περίμενα όμως να μας επιφυλάσσετε τόσες πολλές εκπλήξεις θετικές ως επιτοπλίστων. Ε, είναι προφανές ότι έχετε στο ενεργητικό σας μεγάλα επιτεύγματα Πραγματικά είστε σε θέση, είστε ένα, είστε ένα κέντρο που ε, είναι σε θέση να στέκεται στον ανταγωνισμό, σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά όπως αυτή της μετάφρασης. Θέλω να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Σε σχέση με τις μειώσεις προσωπικού, είπατε ότι αφορούν Ε, το προσωπικό κατά κύριο λόγο βεβαίως που επομίζεται όλο και περισσότερη δουλειά ε, έχουμε και μια μείωση του προϋπολογισμού βεβαίως που ενδεχομένως ε, να μην έχει πολλές να μην φανούν οι επιπτώσεις του τόσο βραχυπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα πρέπει λοιπόν να επαγρυπνήσουμε όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις, τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η μείωση της χρηματοδότησης. Ε, τρία είναι τα βασικά θέματα που νομίζω ότι πρέπει να σταθούν στο επίκεντρο της προσοχής μας. Πρώτον, πρέπει να προστατεύσουμε την πολυγλωσία. Την γλωσσική ποικιλομορφία και πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βάση δεδομένων, λοιπόν, πρέπει να, να διευρυνθεί Και να μην ξεχνούμε ότι ορισμένες εθνικές γλώσσες χάνουν λέξεις από το λεξιλόγιο τους, ολόκληρες κατηγορίες πολλές φορές. Είναι λέξεις που θεωρούνται παροχημένες, παλιωμοδίτικες, που παρόλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να καταγράφονται επιστημονικά στις βάσεις δεδομένων ε, για να μην φτωχύνουν οι γλώσσες. Επίσης μειώθηκαν ε, και οι θέσεις πρακτικής άσκησης ε, που υπάρχουν στον ε, οργανισμό σας. Ενώ αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης αποτελούσαν πάντοτε ένα πρώτο βήμα για να μπορεί κανείς, ένας νέος άνθρωπος να εισέλθει στον κλάδο των γλωσσικών επαγγελμάτων. Και νομίζω ότι ε, η παρουσία σας σήμερα εδώ μας δίνει την ευκαιρία να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η πολυγλωσία ε, ε, μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον άλλον ε, και να ανταλλάσσουμε απόψεις αλλά και γνώμες για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε το, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ξέρουμε ότι εσείς ε, δεν ε, έχετε ως καθήκον σας τη διερμηνία αλλά τις μεταφράσεις, αλλά είναι γεγονός σε κάθε περίπτωση ότι η συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων και σε πολύγλωσσο επίπεδο είναι πολύ σημαντική. Άρα εμείς θα πούμε ότι θα, και σας διαβεβαιώνουμε γι' αυτό ότι ε, θα αντιταχθούμε ε, στις μειώσεις, στις περαιτέρω μειώσεις ε, ε, που έχουν σχεδιαστεί. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας αυτή με τα πολύ ενδιαφέροντα και ολοκληρωμένα στοιχεία. Ευχαριστώ η Σαμπίνε Φερχάιεν. Ευχαριστώ και εγώ για τις ε, πληροφορίες αυτές, για τη δουλειά που κάνετε. Έχω όμως ένα ερώτημα. Υπάρχει ε, εξωτερική ανάφηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι μεταφράσεις ανατίθενται σε εξωτερικές εταιρείες ε, και πολύ συχνά προκύπτει το εξή πρόβλημα. Όταν χρησιμοποιείται ως κείμενο πηγή, το αγγλικό κείμενο, κάτι που προκύπτει και από τις, από, από, από τις συνολικές σας δημοσιεύσεις, ε, ότι ε, πολλές φορές τα αγγλικά ε, υπάρχει μια λέξη η οποία μπορεί να αποδοθεί με 10 διαφορετικούς τρόπους σε κάποια άλλη γλώσσα. Πώς εξασφαλίζετε εσείς σε συνεργασία και με τους εξωτερικούς σας παρόχους ότι θα εξασφαλίζετε το σωστό συγκείμενο. Ε, και η σωστή απόδοση, διότι πολλές φορές έχουμε δει να ε, υπάρχουν μεταφραστικά προβλήματα, να διαβιβάζονται τα μηνύματα στις άλλες γλώσσες με λάθος τρόπο, να το πω καθαρά. Ε, πώς, πώς θεσμικά λοιπόν εξασφαλίζετε εσείς το νόημα της κάθε, του κάθε όρου και της κάθε λέξης να αποδίδεται σωστά στη διαδικασία των μεταφράσεων. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Πράγματι και σε εμά έχει συμβεί πολύ συχνά αυτό. Ιδίω όταν γίνονται, πολύ, πολύ, ε, γίνονται συζητήσει ε, ιδιαίτερα τεχνικέ, που δεν είναι πάντοτε πολύ σαφή τα, τα, τα θέματα αυτά και στου ίδιου μεταφραστέ. Ε, οι οποίοι προφανώς δεν είναι δυνατόν να ε, γνωρίζουν τα πάντα σε όλα τα θέματα του επιστητού. Ε, βεβαίως από την άλλη πλευρά ε, η δική τους δουλειά είναι εκείνη που διευκολύνει και τη δική μας δουλειά και κάποιες φορές μόνο ε, δημιουργούνται προβλήματα κατανόησης ή μετάφρασης. Κυρία Κώστα, Σίλβια, έχεις το λόγο. Ναι. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πανοραμική εικόνα που είναι τόσο εμπεριστατωμένη και ενδιαφέρουσα. Είναι πολύ χρήσιμη για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο. Όλοι πρέπει να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτή τη δουλειά σας. Ήδη από πέρσι είχαμε ακούσει διάφορα προβλήματα προπολογισμού και δυσκολίες που αντιμετώπιζε η διεύθυνσή σας ε, ε, λόγω μιας νέας προσέγγισης και σε σχέση με το ίδιο το θέμα της ε, τεχνικής πρόθεσης ε, ε, του προϋπολογισμού είπατε ότι αυτή η δυνατότητα γιατί περιορίζονται οι δαπάνες για όλους τους θεσμούς και για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς θα πρέπει να συνεχιστεί, μπορεί να συνεχιστεί και μετά θα πρέπει να υπάρξει μια αύξηση οπωσδήποτε. Εσείς μου φάνηκε να λέτε ότι αυτός ο ορίζοντας είναι το 2020 και επειδή μιλάμε για το προπολογισμό του Κοινοβουλίου, μου είπατε, θέλω να καταλάβω ποιο, είναι το περιθώριο. Ναι, το 2020 και έπειτα μια ιδιαιτερότητα. Είδα ότι θέλετε να ενεργοποιήσετε νέες υπηρεσίες. Θέλω να καταλάβω καλύτερα ποιες είναι, ποιες είναι αυτές. Ας πούμε, η μετάφραση online, η άμεση και θέλουμε να ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό ποιοτικά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πολύ συχνά οι επιγραμμικές αυτές εκδοχές δεν είναι σωστές και έπειτα αυτές οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι, τα εξωτερικά γραφεία μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα ας πούμε και στην νομική μετάφραση και στην πολιτιστική γιατί βλέπω συχνά στην Ιταλία στα Ιταλικά ας πούμε δεν μεταφράζεται απόλυτα σωστά πάντα είναι πολύ λεπτά εκεί τα νοήματα φαντάζομαι ότι αυτό το κάνετε εσείς έχετε βρει γραφεία ποιοτικά στην αγορά ή όχι η Julie Ward Εγώ θέλω να πω ότι εκτιμώ πολύ τις λεπτομέρειες που μας παρουσιάσατε σήμερα και πραγματικά πιστεύω πως αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να παίξει πρωταθλητικό ρόλο υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δικό μας θέμα και είναι και εντολή της Επιτροπής μας να σεβαστούμε και να προωθήσουμε τη γλωσσική πολυμορφία και διαφορετικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε οι πρωταθλητές στις πολιτικές μας ομάδες και στις διάφορες ε, επιτροπές. Κάτι που με ενδιαφέρει πολύ είναι να δω τον κατάλογο άλλων γλωσσών που είναι εκτός ένωσης, όχι τις επίσημες γλώσσες, αλλά τις άλλες γλώσσες από τις οποίες και προς τις οποίες μεταφράζεται. Ε, δεν νομίζω ότι ο κόσμος το γνωρίζει αυτό πολύ καλά και προφανώς είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη σχέση και τις σχέσεις με άλλες χώρες, ιδιαίτερα Νομίζω έχουμε τη στρατηγική της πολιτιστικής διπλωματίας και την πρωτοβουλία με τη Φεντερίκα Μογερίνη και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να το στηρίξω και εγώ και πραγματικά είναι σπουδαίο που ήρθατε και μας το παρουσιάσατε αυτά σήμερα. Κάτι ακόμα. Ε, υπάρχουν ε, πολλές ευκαιρίες υπάρχουν. Ε, εγώ, εγώ καλώ κόσμο στο γραφείο μου να έρθει να δει πώς δουλεύει το κοινοβούλιο και κάποιοι πραγματικά ήρθαν γιατί ενδιαφέρονται για τις γλώσσες και μπόρεσαν να ε, συναντήσουν και κάποιους από τους διερμηνείς και αυτό τους φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν υπάρχει η δυνατότητα να έρθουν και να επισκεφτούν και να γνωρίσουν και ε, υπαλλήλους του δικού σας κέντρου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα την Κομισιόν αν θέλει και εκείνη να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι οι λόγοι για τους οποίους ο Ευρωπαίος νομοθέτης δημιούργησε αυτό το κέντρο μετάφρασης το 1994 ισχύουν ακόμη και νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το μοντέλο διότι είναι το πιο κοστοποδοτικό μοντέλο η εξασφάλιση της πολυγλωσσίας ε, είναι βεβαίως ζωτική σημασία για κάθε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί με τους Ευρωπαίους πολίτες ενώ όσον αφορά τη, το, τις μειώσεις προσωπικού θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι οι μειώσεις αυτές ε, τίθενται σε διαπραγμάτευση, σε τήσια βάση και ε, συμφωνούνται από τα τρία θεσμικά όργανα, Κοσμισιόν, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ο αριθμός του προσωπικού θα ε, παραμείνει σταθερός από το 2018 και έπειτα. Δεν προβλέπονται δηλαδή μειώσεις του προσωπικού για το 2019 και το 2020. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν, λέει Πρόεδρος, και θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Κίλωραν, προκειμένου να απαντήσει σε αυτή την πλειάδα ερωτήσεων που ακούστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα θέματα που έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις μειώσεις ε, προσωπικού και τις χρηματοδοτικές μειώσεις, ε, είναι πλέον γεγονότα αυτά. Προσπαθούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας πρακτική και ε, σημειώνω ε, αυτό που είπε η Κομισιόν ότι από το 2018 και έπειτα δεν θα υπάρξουν άλλες σημειώσεις προσωπικού κάτι που βεβαίως μας χαροποιεί ιδιαίτερος. Όσον αφορά τις θέσεις πρακτικής άσκησης πράγματι εμείς έχουμε ασκούμενους και εκπαιδευόμενους ε, στην μετάφραση στο κέντρο μας. Όσον αφορά την παρέμβαση της κυρίας Ward, να πω ότι εμείς είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Αν κάποιος θέλει να κάνει αίτηση και να κάνει πρακτική άσκηση, βεβαίως είναι ευπρόσδεκτος. Πολλές ε, θέσεις ε, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας κάθε χρόνο. Όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση, ε, από την αρχή της, ε, από τη δημιουργία του κέντρου μας ε, ήταν πάγια πρακτική μας αυτή και αυτό βλέπετε ότι έχει ως επιχειρησιακό μοντέλο επεκταθεί και σε άλλους οργανισμούς. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα ε, αναθέτουν όλο και περισσότερη δουλειά σε εξωτερικούς συνεργάτες. Για μας το outsourcing είναι συστατικό στοιχείο της δουλειάς μας. Αναθέτουμε μεταφράσεις σε εξωτερικούς παρόχους. Εμείς ε, στη συνέχεια ελέγχουμε την ποιότητα της μετάφρασης. Πώς το κάνουμε αυτό. Ε, οργανώνουμε διαγωνισμούς θεματικούς ε, στους ιδεοδρόμους, στην αεροπορία, στο περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι οι εξωτερικοί μας πάροχοι έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη. Το ίδιο ισχύει και την ορολογία, διότι ε, αν δεν υπάρχει συμφωνηθής ορολογία που θα χρησιμοποιείται στις μεταφράσεις, τότε πράγματι ε, αντιμετωπίζονται και δημιουργούνται πολλά μεταφραστικά προβλήματα, τα οποία στη συνέχεια καλείστε να αντιμετωπίσετε εσείς. Βεβαίως σημαντικό, σημαντική είναι και η ποιότητα των κειμένων πηγή. Αν τα κείμενα πηγή είναι κακά από άποψη ποιότητα, κατά αντιστοιχεία κακές αναγκαστικά θα είναι και οι μεταφράσεις να, να επιβεβαιώσω και εγώ ότι τα αγγλικά είναι η γλώσσα στην οποία λαμβάνουμε τα περισσότερα ε, κείμενα. Πράγματι ισχύει αυτό, αλλά δεν είναι η μοναδική γλώσσα. Εμείς ε, ανταποκρινόμαστε πάντοτε στα αιτήματα των πελατών μας. Αν τα κείμενα που μας στείλουν είναι αγγλικά, από αγγλικά μεταφράζουμε. Όσον αφορά τα το ερώτημα της κυρίας Κώστα για την ε, περίοδο έως το 2020 θα προσπαθήσουμε να ε, διευρύνουμε τις υπηρεσίες μας αλλά και να προσφέρουμε και νέες υπηρεσίες ε, για παράδειγμα μια υπηρεσία μετάφρασης ιστοσελίδων όλοι οι οργανισμοί έχουν ιστοσελίδες πλέον θέλουμε να τους βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε την ε, παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών για τις ε, ε, ιστοσελίδες. Επίσης, το επόμενο διάστημα σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε και ένα σύστημα μηχανικής μετάφρασης σε συνεργασία με την Κομισιόν, το οποίο θα εφαρμόσουμε. Βεβαίως η μηχανική μετάφραση μόνο υποστηρικτικά μπορεί να ε, λειτουργήσει, ε, υποστηρικτικά για τους ε, ανθρώπους μεταφραστές δηλαδή. Μπορούν να μας βοηθήσουν στην επιτάχυνση της δουλειάς και την εξασφάλιση της ποιότητας. Δεν μπορούν οι μηχανές από μόνες τους να αναλάβουν την μετάφραση. Όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα, νομίζω ότι το μοντέλο μας μας έχει βοηθήσει στο να μειώσουμε το κόστος της μετάφρασης, διότι μέσω της, του outsourcing έχουμε μειώσει τον αριθμό των μεταφραστών που ε, απασχολούμε επίσης. Ε, βεβαίως ε, ε, έχουμε εσωτερικούς μεταφραστές οι οποίοι επιφορτίζονται κατά κύριο λόγο με την εξασφάλιση της ποιότητας διότι το να δίναμε τις μεταφράσεις έξω και να τις στέλναμε απευθείας στους πελάτες χωρίς να έχουν περάσει από το δικό μας φίλτρο θα μπορούσε να ενέχει πολλούς κινδύνους για τη μεταφραστική ποιότητα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για τις απαντήσεις σας και για το γεγονός ότι ε, για πρώτη φορά τουλάχιστον ε, στη δική μου παρουσία εδώ στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με, με την Διευθύντρια του Κέντρου, για το οποίο είμαστε κι εμείς ε, ε, αρμόδιοι άλλωστε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το, η σημερινή μας ε, συνάντηση ήταν η απαρχή μιας πολύ καλής σχέσης, μια πολύ καλής συνεργασίας, μια πολύ καλής φιλίας Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτήν την εξαιρετική μας επαφή που ξεκίνησε σήμερα για πρώτη φορά. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για, την, για όλο το, το, το, το έργο σας που μας διευκολύνει στην καθημερινή μας δουλειά διότι χωρίς μετάφραση και των εγγράφων αλλά και χωρίς διερμηνία στη διάρκεια των συνεργάσεων δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς το έργο μας. Η πολυγλωσία λοιπόν αποτελεί υποχρέωση και καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί έκφραση άλλωστε και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας η οποία πρέπει να εξασφαλιστεί, να διασφαλιστεί και να πω επίσης ότι ε, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι η ποιότητα μιας μετάφρασης εξαρτάται πάντοτε από την ποιότητα των κειμένων από τις οποίες έχουν προέλθει. Ίσως αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως έκκληση ε, οι συγητές μας να μην συντάσσουν τις εκθέσεις τους κάθε φορά τουλάχιστον στα αγγλικά. Καλύτερα ενδεχομένως κάποιες φορές να συντάσσουν τις εκθέσεις τους στην μητρική τους γλώσσα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει και εσάς στο δικό σας έργο. Ξέρουμε ότι δεν είναι πάντοτε εφικτό κάτι τέτοιο. Πολλές φορές υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί που οδηγούν τους εσηγητές να αποφασίζουν να συντάξουν την έκθεσή του στα αγγλικά απευθείας γιατί τα πράγματα έτσι θα προχωρήσουν πιο γρήγορα. Παρ' αυτά... Ε, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε, τις περισσότερες φορές ε, ένα κείμενο που έχει συνταχθεί στη μητρική γλώσσα του συντάκτη είναι πάντοτε πιο εύκολο να μεταφραστεί στη συνέχεια από ότι αν πάω εγώ για παράδειγμα να συντάξω ένα κείμενο στα γαλλικά που δεν είναι η μητρική μου γλώσσα όπου και μπορεί να, η ποιότητα του κειμένου αυτού να μην είναι ιδιαίτερος υψηλή. Ε, αυτό κύριε Σδρογεύσκη ε, όπως είπαμε ε, συντάσσεται και μια έκθεση όσον αφορά την απαλλαγή του κέντρου μετάφρασης και νομίζω ότι και στο μέλλον ε, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να μην μειωθούν περαιτέρω οι πόροι που έχετε στη διάθεσή σας. Αν Πάντως, αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ως προς αυτό το θέμα. Ε, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας. Ε, ελπίζω να έχουμε μια συχνή και η καλής ποιότητας επαφή να διαβιβάσετε όλους τους ε, θερμότερους ε, χαιρετισμούς ε, των μελών της Επιτροπής μας σε όλους τους εργαζόμενους του Κέντρου Μετάφρασης και σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσίασή σας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι να ανακτήσουμε λίγο τις δυνάμεις μας. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν. Α, όχι, συγγνώμη. λάθο τα λέω. κάτι ξέχασα. Όχι, δεν, δεν, δεν είστε ελεύθεροι να φύγετε, διότι έχουμε μία ε, συνεδρίαση ε, και κλεισμένο των θερών. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όσοι δεν είναι μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσοι δεν είναι βοηθοί ευρωβουλευτών, να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Αυτό ισχύει και για τους εκπροσώπους